Καθίστε στις θέσεις σας παρακαλώ, ξεκινάμε. Parlano. Non vogliono sedersi. Sit down, no. Sit down, please. καθίστε παρακαλώ. Ωραία. Καλωσορίζουμε τον κύριο Άιλετ. Είμαστε στην πέμπτη ακρόαση για την θέση του διευθυντή της Όλαφ. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Όπως έγινε και με τους άλλους υποψήφιους, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ο κύριος Άιλετ έχει στη διάθεσή του πέντε λεπτά για να κάνει την παρουσίασή του. Μετά θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις των συναδέλφων ανάλογα με τη σειρά που είχε αποφασιστεί. Κύριε Άιλετ, Νίκ, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι δεν θα πρέπει να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Πολύ, πολλά από τα μέλη της Επιτροπής μιλάνε αγγλικά και δεν ήθελα να σας απευθυνθώ στα αγγλικά για να μπορέσει να περάσει το αρχικό μου μήνυμα. Μετά θα μιλήσω και σε άλλες γλώσσες. Εκτό Εκτός από τη γραπτή μου ομιλία θα ήθελα τρεις παρατηρήσεις να κάνω. Πρώτα απ' όλα σχετικά με την ΟΛΑΦ. Η ΟΛΑΦ έχει δύο ρίζες. Μία οικονομική από τον προπολογισμό και μία δικαστική από την επιβολή του νόμου. Εγώ ήρθα στην ΟΛΑΦ από τον οικονομικό κλάδο. Η ΟΛΑΦ είναι μια υπηρεσία καταπολέμησης απάτης 360 μοιρών. Αντιμετωπίσει όλο τον κύκλο καταπολέμησης απάτης από την διακρύβωση των στοιχείων, την συγκέντρωση πληροφοριών, την ανάλυση, καλύτερη πρόληψη, διαμόρφωση πολιτικής και νομοθεσία. Η ΟΛΑΦ πρέπει να διατηρήσει όλες αυτές τις αρμοδιότητες. Η ΟΛΑΦ είναι μοναδική δεν μπορείτε να πάρετε ένα μοντέλο από κάπου αλλού, να το πετάξετε στην περιοχή που υπάρχουν τα κτίρια τα ευρωπαϊκά στην Ευρώπη και να περιμένετε ότι θα λειτουργήσει. Η ανεξαρτησία της Όλαφ από άποψη είναι αποφασιστική σημασία για την Όλαφ, η οποία είναι ένας πυλώνας εμπιστοσύνη. Εγώ θα μεριμνήσω να υπάρχει αυτή η ανεξαρτησία, ό,τι και αν συμβεί. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι ότι τα, τα επόμενα πέντε χρόνια η Όλαφ θα αντιμετωπίσει θεσμικές προκλήσει, αλλά και διαχειριστικέ προκλήσεις. Οι θεσμικές προκλήσεις συνίστανται στο να εφαρμόσει την παρούσα μεταρρύθμιση της Όλαφ και κατόπιν να καταστεί ικανή να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας όπως αποφασίσει ο νομοθέτης. Ελπίζεται ότι η Όλαφ θα παίξει σημαντικό ρόλο ως διοικητικός φορέας για να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Σαγγελική Αρχή. Το άμεσο έργο του Γενικού Διευθυντή είναι να φροντίσει να λειτουργήσει η μεταρρύθμιση χωρί να αυξηθεί η γραφειοκρατία, κυρίως όσον αφορά τα ατομικά δικαιώματα. Όπου παρεμπιπτόντω υπάρχει φόβο οι αξιωματούχοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε άλλον, λάθο επιλογή θα έλεγα. Είναι ουσιαστικό η μεταρρύθμιση να διευκρινίσει την διακυβέρνηση Όλαφ. Θα πρέπει να καταστεί ο ρόλος της Επιτροπής Εποπτείας ε, λιγότερο συγκεχημένος. Θα πρέπει να λαμβάνονται στρατηγικές αποφάσεις για την κατανομή των πόρων. Μεταξύ αφενός, για παράδειγμα, μεγιστοποίηση του οικονομικού αντίκτυπου της δραστηριότητα της Όλαφ ή τη μεγιστοποίηση της γνώσης των άλλων για την Όλαφ. Δηλαδή προστασία των εισοδημάτων και καταπολέμηση διαφθοράς ή μεταξύ έρευνα και και πρόληψης. πρωτοβουλίες και όχι ένα στρατηγικό σχέδιο. Θα επαναθεωρήσω τις προτεραιότητες, της στρατηγικές της Όλαφ, θα συμβουλευτώ τους εμπλεκομένους, συμπεριλαμβανομένης και της Επιτροπής, θα αναδιοργανώσω, θα επαναισορροπήσω και θα εστιάσω και πάλι στις δραστηριότητε τη Όλαφ για να αντιμετωπίσω τις αλλαγέ που αντιμετωπίζει η Όλαφ. Η Όλαφ πρέπει να προσθέσει αξίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο με την κεντρική της θέση και το προσωπικό με πολλαπλές γνώσεις που αντιπροσωπεύει πολλές κουλτούρες. Θα πρέπει να εστιάζεται στους πιο σημαντικού κινδύνους από την πρόσφατη, τη μελλοντική διεύρυνση στο οργανωμένο έγκλημα, στα ανατολικά σύνορα και στα μεγάλα προγράμματα δαπανών που θα πρέπει να προστατεύει. Αυτό απαιτεί κάποια αναδιοργάνωση και ανακατανομή των πόρων, αλλά απαιτεί επίσης ορισμένες δύσκολες αποφάσεις. Τέλος, έρχομαι στην προσωπική μου εμπειρία στον τομέα των ερευνών. Ποτέ δεν υπήρξα ένα άτομο που δούλευε έξω. Αντιμετώπισα τους νέους ε, με περίπλοκα οικονομικά θέματα για παράδειγμα ανταλλαγή πληροφοριών για την αντιμετώπιση της απάτης, ε, ε, κυρώσεις για φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή κτλ. Θα πρέπει και η διαγνωτική διαδικασία στην Όλαφ να το ακολουθεί, ώστε ε, να προχωρήσει Όλαφ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα γερμανικό κείμενο, το οποίο απαιτεί στην αίτηση υποψηφιότητων απαιτεί. σε μια ηγετική θέση, σε, μια, σε ένα κράτος μέλος μιας παρόμοιας υπηρεσίας. I have been in precisely such a position in OLAF for nine years and in four roles, as Director for Intelligence, then Director for Policy, and in the last nine months as Acting Director General. Thank you. Grazie Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις με την κυρία Γκρέσ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χάιλετ. Γνωριζόμαστε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Η ερώτηση που θα διατυπώσω δεν θα σας εκπλήξει βέβαια. Η μεταρρύθμιση της Όλαφ είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει ως κύριο θέμα τα επόμενα χρόνια και σίγουρα θα το προτιμούσα αν σε αυτό το σημείο είχαμε προχωρήσει πιο πέρα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, χωρί τη την υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή τη Όλαφ, αυτή η μεταρρύθμιση δεν θα μπορέσει να, να γίνει. Έχω τώρα σε ανάμνηση την παρουσίαση της ε, εισήγησης. Είχαν παρουσιαστεί σοβαρές επικρίσεις ε, και ξέρω ότι η δική σας γνωμοδότηση έτυχε μιας αρνητικής παρατήρησης από πλευράς γραμματέως. Είσαστε τότε αναπληρωτής, δεν μπορούσατε να πάτε πιο πέρα. Ερώτηση. Αυτό το γεγονός είναι πραγματικά κάτι που έχω δραματικά ακόμα στη μνήμη μου και γι' αυτό θα ήθελα να θέσω το ερώτημα. Πόσο ανεξάρτητος είσαστε πραγματικά και πόσο ανεξάρτητος θα είσαστε πραγματικά και ποια είναι η δική σας θέση σε σχέση με ε, την ε, προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τέτοιες προτάσεις μεταρρύθμισης όπως από την πλευρά. Θα ήθελα κυρία Γκρέσλε αυτή τη συζήτηση να την είχαμε κάνει πριν από αρκετό χρονικό διάστημα μαζί σας. Και για μένα ήταν ένα πολύ σοβαρό γεγονός αυτό και έχετε δίκιο σε αυτό. Έχω συνηθίσει όταν μου δίνουν εντολές ως υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπακούω σε αυτές τις επισημάνσεις και κατευθύνσεις και ως Γενικός Διευθυντής όταν και αν εργάζομαι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον πολιτικό ε, στο πολιτικό σκέλος, όχι στο λειτουργικό στις, στη δράση, αλλά στο πολιτικό επίπεδο, τότε είναι αυτονόητο ότι πρέπει να δουλεύω και να εργάζομαι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτή ήταν η περίπτωση και με τον κύριο Γκρόνερ. Όμως, ανεξαρτησία τώρα στον τομέα των λειτουργικών δράσεων, και των εξεταστικών δράσεων. Αυτό είναι τεράστια σημασία θέμα η ανεξαρτησία. Είμαι ανεξάρτητος και θα παραμείνω ανεξάρτητος. Είμαι ανεξάρτητος, independent και θα παραμείνω independent, ανεξάρτητος, το τονίζω. Με τη μεταρρύθμιση τώρα. Χαιρετίζω αυτή τη μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση είναι αναγκαία. Χρειαζόμαστε σαφείς ενδείξεις χρειαζόμαστε σαφή και καθαρή διαχείριση και διακυβέρνηση, μεγαλύτερη αποσαφήνιση για τα δικαιώματα. Υπάρχουν διεργασίε, διαδικασίες που πρέπει να βελτιωθούν. Υπάρχουν αδυναμίες ε, στην αρχική νομοθετική πρόταση που πρέπει να επανορθωθούν. Υποστηρίζω πλήρω αυτό το στοιχείο για τη μεταρρύθμιση και θα εργαστώ όταν και αν θα είμαι Γενικό Διευθυντή για να υλοποιηθούν αυτά. Πρώτον, επικοδομητικά στη φάση των συζητήσεων και διαβουλεύσεων ως υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά επίσης εκπροσωπώντας και τις επαγγελματικές απόψεις της Όλαφ που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη μεταρρύθμιση γιατί διαφορετικά αν γίνει κάτι άλλο δεν θα επιτυγχανόταν η μεταρρύθμιση και η νομοθεσία δεν θα ήταν ιδανική. Και πάλι επίσης όπως αναφέρω στη γραπτή μου δήλωση ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνω στο να εφαρμοστεί οι μεταρρυθμίσεις σε όλες τις λεπτομέρειες όταν θα έχει προχωρήσει αυτή. Ζητώ συγγνώμη αν ε, χρονοβόρησα. Ε, Γκάιερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Χάιλετ, προσέξτε. Ας ξεκινήσω διαφορετικά. Την ερώτηση ήδη στην παρουσίαση της ε, ε, έκθεσης, ε, γενικής έκθεσης για το έτος την είχα διατυπώσει. Ας αντιμετωπίσω το θέμα διαφορετικά. Δεν είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την κατάσταση ότι ο αριθμός όσων εργάζονται για έρευνες στην Όλαφ είναι περίπου, κάτω από ένα, περίπου στο 1 τρίτο. Όλοι οι υποψήφοι που ακούσαμε μέχρι τώρα στην παρουσίασή τους συμφωνούσαν όλοι ότι αυτή η αναλογία, αριθμητική αναλογία πρέπει να αλλάξει πλέον. Τώρα, Βλέποντας το οργανωτικό ε, πρόγραμμα της Όλαφ, αν το θυμάμαι καλά, εσείς προτού γίνετε διάδοχος του κυρίου Γκρόνερ, είσαστε Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας ΔΕΛΤΑ. Δηλαδή, δεν το αναφέρω με τέλειο τρόπο τώρα, τυπικά, ως τον τίτλο, είσαστε αρμόδιος για την προετοιμασία των στοιχείων για τις ερευνητικές δραστηριότητες. Αν γίνεται όμως ε, Γενικός Διευθυντής της Όλαφ, θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας ε, ο αριθμός των στελεχών να αυξηθεί. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει την αποδυνάμωση εντός εισαγωγικών της παλαιάς ε, διευθυντικής σας θέσης και του τομέα που είχατε πριν εσείς στην εξουσία. Αυτό δεν αφορά το μέγεθος της διεύθυνσης το μεγαλύτερο μέρος της διεύθυνσης ασχολείται με την ε, πληροφορική και την διαχείριση πληροφοριών από πλευράς των ερευνητών. Αλλά είμαστε και ένα έρισμα για τις ε, τελωνιακές υπηρεσίες. Αυτό είναι μέρος της εργασίας μας του συντονιστικού ρόλου δηλαδή που παίζει όλα. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ερευνητών, αλλά η άμεση προτεραιότητα για μένα είναι, ε, έχει σχέση με το θέμα της ε, πληροφόρησης και το θέμα των ε, αναλυτών ιατροδικαστικής. Το θέμα είναι να μπορέσει η πραγματογνωμοσύνη αυτή να συμβάλλει στο να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν άλλοι. Αυτό συνεπάγεται την αύξηση του προσωπικού της διεύθυνσης. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να ενδυναμωθεί. Το επόμενο ερώτημα είναι πού θα βρούμε αυτό το προσωπικό. Δεν μπορώ να κλείσω το πολιτικό κομμάτι, το, κομμάτι της πολιτικής της όλα. Χρειάζεται χρειάζονται άνθρωποι για να ασχολούνται με το θέμα της πολιτικής της Όλαφ. Εάν σταματήσουμε να χαράσουμε πολιτική, θα μπορούσαμε να διοχετεύσουμε περισσότερους ανθρώπους στον τομέα της έρευνας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περικοπές στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, ενδεχομένως Έξι, επτά, 8 άτομα θα μπορούσαν να ασχοληθούν με περισσότερο λειτουργικό έργο. Τα τελευταία δύο χρόνια μείωσα τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της πολιτικής. Με τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου Μπούνες ε, διοχέτευσα μερικούς από αυτούς τους πόρους στην ε, έρευνα και άλλους στην πληροφόρηση. Για να γίνει όμως μια πιο ε, διαφορά θα πρέπει να αλλάξουν άλλες λειτουργίες της όλα. Θα πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε κάτι που κάνουμε τώρα. Και αν μεταφέρουμε ε, ορισμένες θέσεις σε άλλες διευθύνσεις θα γίνει αυτόματη μεταφορά των πόρων. Ας πούμε, ε, όπου μεταφερθεί η προστασία θα μεταφερθούν και οι ε, πόροι προστασίας. Ο συνάδελφος Τάις ζήτησε να του δοθεί ο λόγος νωρίτερα γιατί θα πρέπει να πάει σε μια επιτροπή. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ που αλλάξατε την διάταξη, αλλά είμαι συγητή σε μια επιτροπή και πρέπει να ψηφίσω, λοιπόν θα πρέπει να αποχωρήσω σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Ζητώ συγγνώμη και στο δύο Λέτα, αλλά κάποιο θα με ενημερώσει σχετικά με τόσα υπόθηκαν. Γνωρίζετε ίσως τι ερώτηση θα σας κάνω, διότι αυτό το ερώτημα το έκανε και στον κύριο Κρετά στις επαφές που έχουμε με τα μέλη και τους συνεργάτες ΟΛΑΦ. Συχνά έχω την εντύπωση ότι στα πλαίσια των υπηρεσιών υπάρχουν ορισμένε συγκρούσεις. Μάλιστα γίνεται λόγος και για δημιουργία ορισμένων ομάδων. Ε, το ερώτημά μου είναι το εξή. Έχετε επίγνωση αυτού του προβλήματο. Είναι αληθές και αν ναι, ποια είναι τα μέτρα που επιθυμείτε να λάβετε ως Γενικό Διευθυντής για να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Euh, κύριε Πρόεδρε, κύριε Στάση, ζητώ συγγνώμη καταρχήν. Διότι όταν έγινα Γενικό Διευθυντής ε, ήμουν υποχρεωμένος ε, για λόγους φόρτου εργασία τη ε, μελέτη μου των Ολλανδικών. Γι' αυτό δεν θα σας απαντήσω στη γλώσσα σας. Γεγονός είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει εδώ και καιρό. Ε, φέρουμε ένα βάρος του παρελθόντος, το οποίο κουβαλάμε μαζί μας. Η κατάσταση λοιπόν δεν είναι όμως και τόσο κακή όπως λέγεται. Η πλειοψηφία, στην εθνική πλειοψηφία των συναδέλφων θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εκείνοι που έρχονται να σας δουν και ίσως και οι συνάδελφοι που έρχονται να επισκεφθούν ορισμένους συναδέλφους σας είναι εκείνοι που δεν είναι ευτυχείς, αλλά αυτή είναι η μειοψηφία, η μειονότητα και έχουν ορισμένα να ρυθμίσουν, ε, έχουν τους δικούς λογαριασμούς. Δηλαδή, το σκέφτηκα πολύ αυτό το θέμα και κατέληξα στο εξή συμπέρασμα. Το πρώτο, όταν ε, προσλαμβάνουμε πολλούς συναδέλφους που έρχονται από την, ε, τις δυνάμεις καταστολής, ε, τις δυνάμει, ε, δυνάμεις, είναι πιο σκληροί, όπως λέμε. Δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Δεν πιστεύουν πάντοτε αυτά που τους λέμε ή που τους λέω. Συνεπώς αυτά τα άτομα έχουν χαρακτηριστικά διαφορετικά. Είναι διαφορετική. Είναι άτομα που τα χρειαζόμαστε για τη δουλειά μα. Και είναι διαφορετικό από την Επιτροπή. Είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσει κανεί αυτά τα άτομα. Γι' αυτό το λόγο είναι ο χαρακτήρα του. Είναι η κατάρτισή του, η εκπαίδευσή του αυτή. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Εάν πιστεύετε ότι έχουμε προβλήματα στην Όλαφ, καλύτερα να κοιτάξετε τι υπηρεσίε των άλλων διεθνών οργανισμών τον ΟΗΕ, την Παγκόσμια Τράπεζα, όπου τα προβλήματα είναι πολύ χειρότερα, ειλικρινά. Και φοβούμε ότι αυτά χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες γενικά, τις μεγάλες υπηρεσίες. Τώρα, η διαδικασία ενσωμάτωσης των προσωρινά εργαζόμενων. Ε, είναι ένα θέμα δύσκολο και θα το έχουμε και αυτό στην πλάτη μας. Αλλά θα πρέπει και αυτό να το λύσουμε. Τρίτο, το μέσα στο προσωπικό της Επιτροπής υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των βαθμών και των μισθών ατόμων που επιτελούν το ίδιο έργο. Και αυτό δημιουργεί και ζήλες και δυσκολίες στη διοίκηση. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Εγώ τα, τα βλέπω με, με την επικοινωνία που έχουμε. Όταν ρυθμιστεί η διαδικασία μας τα πράγματα θα διευκολυθούν. Αλλά συμφωνώ μαζί σας, είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών είναι πολύ σημαντικό. Σε ποιου τομεί ε, θα βελτιώσετε την ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη-μέλη, κυρίω πώς μπορείτε να φροντίσετε ότι θα υπάρχει καλύτερη δικαστική παρακολούθηση όλων των υποθέσεων. Ευχαριστώ. Η επικοινωνία με τα κράτη-μέλη ε, γίνεται σε πολλά επίπεδα και διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα και ανάλογα με την υπηρεσία στην οποία απευθυνόμαστε σε ένα κράτο μέλος. Μπορώ να ε, τηλεφωνήσω στο, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και να τον δώσω σε δύο μέρες. Εάν τηλεφωνήσω στο δικό μου Πρωθυπουργό θα δω έναν Υφυπουργό ίσως σε δύο μήνες. Αυτό εξαρτάται από τις περιστάσεις και πρέπει λοιπόν να προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας στην κάθε περίπτωση. Τώρα, για τη δικαστική παρακολούθηση. Οι απευθείας επαφές μεταξύ των ειδικών του δικαστικού σώματος και των ειδικών του δικαστικού σώματος των κρατών μελών είναι απαραίτητη. Και όταν είχαμε σε επαφή με Έλληνες δικαστές, οι Έλληνες έκαναν άλμα από το τίποτα σε μεγάλη επιτυχία το να μετρήσει κανείς τη δικαστική επιτυχία είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες εκεί. Τα πράγματα δεν είναι τόσο κακά όπως λέγεται συχνά. Αν δείτε ένα χρονικό ορίζοντα αρκετά μακρινό, θα δείτε τα πράγματα. Αν δείτε ένα μικρό χρονικό ορίζοντα, θα έχετε αυτό το 70% το οποίο είπαμε. Αλλά αν πάρετε ένα μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, αν έχετε μικρό ορίζοντα έχουμε 7%, αν έχετε μεγάλο χρονικό ορίζοντα έχετε 28% περίπου. Δεν μπορώ να σα δώσω πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Πάλι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα ταχύτητας. Το σημαντικότερο είναι, νομίζω, να πείσετε τις υπηρεσίες των κρατών μελών ότι είναι ανάγκη να συνεργαστούν μαζί μας και ότι μπορούν και αυτές οι υπηρεσίες να ωφεληθούν από αυτή τη συνεργασία. Και είναι αυτό προφανέ με ενα κρατη κράτη-μέλη. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Σε άλλα κράτη-μέλη, η σχέση μας είναι ένας εικονικός κύκλος, θα έλεγα. Το καλύτερο παράδειγμα είναι ε, ε, με συγχωρείτε, ένας ενάρετος κύκλος θα έλεγα. Στην Ιταλία υπάρχουν πολύ ικανοί συνεργάτες. Υπάρχει ένας ε, ε, κύκλος εναρέτων ανθρώπων οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μας, αλλά επίσης συμβαίνει και το αντίθετο σε ορισμένα μεγάλα κράτη-μέλη. Αλλά είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά να λειτουργήσουν άψογα. Ο διάβολος βρίσκεται, στα, όπως λέμε, σε λεπτομέρειες και πρέπει να δούμε την κάθε λεπτομέρεια και την αξιοποιήσουμε. Συνάδελφος Μπάρσουντης. Η σημαντική σας εμπειρία στα πλαίσια της ΟΛΑΦ μας ε, καθησυχάζει, αλλά οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες αναφέραμε σήμερα απαιτούν ορισμένες αλλαγές. Το ερώτημά μου λοιπόν μοιάζει με, εκείνο που, με εκείνα που σας τέθηκαν προηγουμένως. Δηλαδή, πώς επικοινωνείτε με τα κράτη-μέλη σε περίπτωση όπου υπάρχει διαφθορά ή απάτη. Σύμφωνα με την έκθεση του 2009, 111 κοινοποίησεις σχετικές ελήφθησαν και οι 94 αφορούσαν τη Βουλγαρία και οι υπόλοιπε τα άλλα κράτη-μέλη. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι, εδώ πρόκειται για έλλειψη ελέγχου από πλευράς κρατών μελών ή δεν λείπει σωστό σύστημα επικοινωνία. Λείπει το σωστό σύστημα επικοινωνία. για να υπάρχουν σωστέ σχέσει μεταξύ τη ΟΛΑΦ και των κρατών μελών. Yes, Ευχαριστώ. Πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα ε, στην ε, κοινοποίηση και τις ε, ατασταλίες στον αγροτικό τομέα, που είναι μια ε, απέτηση η οικονομική διαχείριση. Πολύ σημαντικά στοιχεία για να κάνουμε αναλύσεις και να έχουμε πληροφορίες. Αφενός και την κοινοποίηση στην ΟΛΑΦ συγκεκριμένων ισχυρισμών που έχουν σχέση με πιθανές συγκεκριμένες παρατυπίες και απάτες. Αυτό το οποίο ονομάζουν οι Γάλλοι προσεντήρ ponctuelles, συγκεκριμένες διαδικασίες, όταν υπάρχει συγκεκριμένη ε, παρατυπία ή απάτη. Λοιπόν, το κλασικό δίλημα είναι πώς να κάνει κανείς διάκριση μεταξύ των δύο. Όταν ε, υπάρχουν πολύ λίγες κοινοποιήσεις επειδή η διοίκηση είναι πολυ λιγες κοινοποιήσει, επειδη η διοικηση ειναι θαυμασια και δεν υπάρχουν ατασταλείς ή παρατυπίες ή επειδή η διοίκηση είναι ανίκανη και δεν αποκαλύπτει την αλήθεια. Αυτό είναι το δύσκολο. Να δούμε ε, πού βρίσκεται η αλήθεια. Ουσιαστικά εγώ πιστεύω ότι πολύ λίγες παρατυπίες αναφέρονται σε σχέση με τις δαπάνες σε αυτή τη χώρα. Το οποίο σημαίνει ότι δεν γίνονται αρκετοί έλεγχοι ή ότι δεν μας ενημερώνουν για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Βεβαίως, στην ε, πληροφορίες που πηγαίνουν από τη Γερμανία στο Ξεμούρο δεν αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι πού πηγαίνουν οι δαπάνες ανά πρόγραμμα, ανά έτος, σε κάθε κράτος μέλος και αν κάνετε αυτή την αναλυτική δουλειά τότε θα έχετε αποτελέσματα που θα σας εκπλήξουν και που είναι αρκετά αντιφατικά. Αλλά επανερχόμενοι όμως το θέμα, έχουμε αρκετούς ερευνητές, αυτό είναι ένα έργο που απαιτεί ε, πάρα πολύ πληροφόρηση που διαθέτει αυτή τη στιγμή η ΟΛΑΦ και θα ήθελα να διατηρήσω αυτό το σκέλος της πληροφόρησης. Το βρίσκω πολύ καλά πως ε, εσείς αντιμετωπίζετε αυτό το έργο. Θέλω να επανέλθω στην ερώτησή σας. μετά από τα εσωτερικά προβλήματα, εσείς τοποθετηθήκατε επ' αυτών. Όμως ερωτώ σε Ευρωβουλευτής, αν σε έναν εκπρόσωπο αυτών των οικογενειών ή αυτών των κλάν, δώσω την ψήφο μου, πώς αντιμετωπίζει την άλλη πλευρά, την αντίπερα όχθη. Με ενδιαφέρει αυτό. Διοικητικές υπηρεσίες είχατε εσείς ε, αναλάβει. Παρ' όλα αυτά είναι ένα μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τουλάχιστον αυτό νομίζουμε. Με ενδιαφέρει πώς με την αντίπερα όχθη θα αντιμετωπίζατε εκείνους πώς στους ιτημένους, ας το πω έτσι, θα δίνατε την ευκαιρία να ενταχθούν. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, με όλο το σεβασμό δεν δέχομαι την ουσία της ερώτησης γιατί δεν θεωρώ ότι εκπροσωπώ κάποια φράξια ή κάποια ομάδα από φράξες. Το αποτέλεσμα αυτής τη διαδικασία δεν είναι ότι κάποιος θα είναι υπό σε σχέση με κάποιους άλλους. Εγώ θα στηρίξω οποιονδήποτε οριστεί γενικό διευθυντής και είμαι σίγουρο ότι και άλλοι υποψήφοι θα κάνουν ακριβώς το ίδιο. Έχω την εντύπωση ότι όταν καθήκον σας είναι να συντονίσετε διάφορους τομείς θα πρέπει να καταφέρετε να κάνετε όλους να αποδώσουν εξίσου καλά. Θα πρέπει να καθοριστούν προτεραιότητες βεβαίως. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα όλο όσο περισσότερα συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Ένα από τα πράγματα που είπα στο προσωπικό πέρσι όταν συζητήθηκε αυτό το θέμα είναι ότι ένα μέρος του προβλήματος έγινε στο ότι συμβιώσαμε σε αυτό το κλειστό περιβάλλον για ένα εκτενές χρονικό διάστημα και έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε στις αδυναμίες και όχι στα δυνατά σημεία του καθενός μας. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε την αριστεία, δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για άλλους, την αριστεία που οδήγησε στον διορισμό των ανθρώπων αυτών. Αυτό είπα στην ε, συνάντηση που είχαμε ε, πριν από ε, ένα χρόνο όταν προείδραψα αυτή τη συνεδρίαση. Και νομίζω ότι αυτό έγινε γενικά αποδεκτό. Ε, ακούστηκαν κάτι γελιότητες στις Βρυξέλλες ε, σε μια, μια περίεργη στο σελίδα σε μια χώρα μέλος. Αλλά πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν μεγεθυνθεί. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι της κλίμακας που καριγράφετε εσείς. Θα πρέπει να φανώ σκληρός με ορισμένους ανθρώπους. Και το αν έχετε κάποια επαφή, σας ήρθα σε επαφή μαζί σας, δεν το ξέρω. Αλλά είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί και πρέπει να συνεργαστούμε όλοι από κοινού. Ανδρέας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ράιλετ, Είπατε ότι η Όλαφ είναι υπεύθυνη για τον όλο κύκλο της καταπολέμησης της απάτης. Δεν άκουσα να λέτε πολλά για την ανείχνευση και για την πρόληψη. Τι πρωτοβουλίε έχετε σκοπό να λάβετε για να ενδυναμώσετε τον τομέα τη πρόληψη και τη ανείχνευση. Δεύτερη ερώτηση, τι μεταρρυθμίσει θα προωθήσετε έτσι ώστε να εκμεταλλευτείτε περισσότερο τις πληροφορίες που διάφοροι πληροφοριοδότες θα μπορούσαν να σας δώσουν. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ανείχνευσης, υπάρχουν δύο τρόποι ο ένα τρόπο είναι να περιμένει κανείς να φτάσουν οι πληροφορίες από τους πληροφοριοδότες κυρίως από τις υπηρεσίες της ε, Επιτροπής και από άλλες πηγές. Ο δεύτερος τρόπο είναι να αναζητήσουμε εμεί ε, τις πληροφορίες μέσω της ανάλυσης ιδιαίτερα. Και μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα δίκτυα προέκυψαν από τους μηχανισμούς ανάλυσης. Γι' αυτό αυτό απαιτείται με ένα χειρισμό των στοιχείων για να μπορέσουμε να βρούμε ύποπτους εταίρους. Αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε όταν ήμουν διευθυντής του Τμήματος Πληροφοριών. Στην αρχή οι μεγάλες ε, επιτυχίες προέκυψαν καθώς άρχισαν να έρχονται μαζικά τα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορέσει να λειτουργήσει η υπηρεσία. Αυτή είναι η ανείχνευση. Πρόληψη τώρα. Η πρόληψη σημαίνει ότι μαθαίνει κανείς, ε, από τα, διδάσκεται από το παρελθόν. Έχουμε υποβάλει ε, ορισμένες προτάσεις στην Επιτροπή σχετικά με το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις απάτες. Ε, σε εκτενέστερο επίπεδο κάναμε προτάσεις για άλλου είδου δημοσιονομικέ απάτες ε, για επιχορηγήσεις ε, που δεν αφορούν συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά όλο τον προπολογισμό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ των δύο. Συμβάλαμε και σε συζητήσεις στα πλαίσια της Επιτροπής ε, κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας για, την, ε, για μια νομοθεσία που δεν θα προσφέρεται, δεν θα ευνοεί τις ε, απάτες. Και αυτό είναι κάτι που κάνουμε διαρκώς. Αυτό γίνεται από άτομα που δεν είναι ερευνητέ. Εάν μετατεθούν στον τομέα της έρευνας, ε, θα αμπληθεί η διαδικασία εκεί. Τώρα, οι πληροφοριοδιώτες Κοιτάξτε, αυτό είναι μία διασφάλιση για ένα αποτελεσματικό διοικητικό σύστημα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προφυλάξουμε τις πληροφοριοδέτες. Βεβαίως αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε κανείς να καταχραστεί. Ενδεχομένως θα μπορούσαν να υπάρξουν ε, και περιπτώσεις κακοήθειας. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αφού προηγουμένως το ανοιχνεύσουμε. Έχουμε ένα σύστημα που βασίζεται στην ε, ε πληροφορική, δεν, έχει δεν το έχουμε πλήρως εκμεταλλευτεί. Δυστυχώς, συγγνώμη, ξέρω ότι με πιέζει ο χρόνος. Η ουσία είναι ότι είναι σημαντικό να υπάρχει το σύστημα και να μπορεί να χρησιμοποιείται. Ε, το θέμα είναι ότι υπάρχει το σύστημα. κυρία ε, κυρία Γκρέσλε, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για τι γλωσσικέ σα γνώσει. Σίγουρα είσαστε ο πιο πολύγλωσσος υποψήφιο που είχαμε. Σε ένα πράγμα θέλω να δώσω συνέχεια που αναφέρατε, τον αριθμό δηλαδή των εξεταστικών ε, περιπτώσεων των εξετάσεων. Αν εσεί ε, απελευθερώσετε από τη Γενική Διεύθυνση άτομα γι' αυτό, τότε το συμπέρασμα είναι γιατί δεν έγινε αυτό εδώ και πολύ χρονικό διάστημα προπολού υπάρχουν αντιστασει για την απελευθέρωση προσωπικού και εδώ υπάρχει υπόθεση ότι υπάρχει κάποια τέτοια αντίσταση ώστε να μην χρησιμοποιούνται περισσότεροι για ερευνητικές δραστηριότητες. Θα ήθελα μια δεύτερη ερώτηση να διατυπώσω που αφορά την τωρινή σας δραστηριότητα το θέμα δηλαδή της διοίκησης, της διαχείρισης του Όλαφ. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους προσωρινά απασχολούμενους, με τους συμβατικά απασχολούμενους, προσωρινά δηλαδή απασχολούμενοι. Μια διαρκής λύση πρέπει να εξευρεθεί και αυτό είναι μια προσπάθεια που κρατάει πολύ χρόνο τώρα. Το ερώτημα είναι γιατί παίρνει τόσο μεγάλο χρόνο. Γιατί αυτά τα θέματα δεν έτυχαν μεγαλύτερης προσοχής από εσά και δεν προόδευσαν πιο πολύ. Ευχαριστώ άτομα από τη δική μου διεύθυνση έχω ήδη δώσει στι υπηρεσίε. Ο κύριο Γκρένερ μου είπε ότι υπερβολικά απελευθέρωσα τέτοια άτομα και διέθεσα τέτοια άτομα. Δεν έπρεπε να το κάνω, λέει, πιο πολύ. Διότι εδώ είναι θέμα και πολιτικής ε, που πρέπει να προσέξουμε. Και από τη γενική μου διεύθυνση υπάρχουν υπηρεσίες που είναι, πιο είναι σημαντικές, όλο και πιο σημαντικές. Προστασία προσωπικών δεδομένων, πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες απαντήσεις σας στις ερωτήσεις σας για παράδειγμα εδώ έχουμε δύο διευθύνσει που ασχολούνται και είναι καλέ οι ερωτήσει αυτού του Κοινοβουλίου. Αφορώ, αναφέρομαι σε αυτό το Κοινοβούλιο, σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Και η νομική εργασία, το νομοθετικό πλαίσιο είναι όλο και πιο σημαντικό. Η συνεργασία με τον Ombudsman είναι σημαντική υπόθεση. Χρειαζόμαστε τέτοιε θέσει στη δική μου διεύθυνση. Θα μπορούσα άτομα από τον τομέα τη πληροφοριακή να χρησιμοποιήσω, διότι έχουμε αναπτύξει περισσότερα συστήματα και καλύτερα συστήματα Απάντησή μου σε αυτό το ερώτημα. Έχω ήδη απελευθερώσει και διαθέσει τέτοια άτομα, τέτοια στελέχη. Και είμαι γενναιόδωρο, generous, το έχω κάνει αυτό. Τώρα, για τους συμβατικά απασχολούμενου, προσωρινά απασχολούμενους, επισυμβάσει. Εγώ ίδιο αυτό το πρόβλημα το αντιμετώπισα προ επίλυση μόλις έγινα Γενικός διευθυντή Δυναμικού ε, Στελεχών σε αυτόν τον τομέα μεγάλες δυσκολίες ε, υπήρξαν από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της διοίκησης, αλλά και από πλευράς των συνδικάτων, μεγάλες αντιστάσεις. Όταν ήθελα να ε, καταλήξω σε μια συμφωνία, σε μια σύμβαση μαζί τους, ώστε οι προσωρινά απασχολούμενοι επί συμβάση να γίνουν ε, συμβάσεις αορίστου χρόνου. Και εγώ είμαι, είχα τέτοια σύμβαση προσωρινής απασχόλησης. Είμαι υπερήφανος πρέπει να πω. Είμαι υπερήφανος ότι επί συμβάση ε, εργάζομαι. Υπάρχουν όμως δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα να μετατρέψουν τις συμβάσεις σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Και αυτοί δυστυχώς πρέπει να αποχωρήσουν. Αλλά είναι 10 ή 12. Τους άλλους 60 θα τους ε, διατηρήσουμε και πολλοί έχουν γίνει ήδη υπάλληλοι. Το πρόβλημα έχει επιληθεί λοιπόν. Υπάρχει ο πόνος ακόμα, το πρόβλημα, ε, ε, ο πόνος από το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά το πρόβλημα λύθηκε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Χάιλετ, για αυτό το νέο, τη νέα ιδιότητα για υποψήφιο που, υποψήφιο που είναι για την Γενική Διεύθυνση, θα ήθελα να το χαιρετήσω. Είπατε ότι έχουν διατηρήσει ή διατηρούν ε, τις ε, σημερινές ε, αυτές οι ιδιότητες τους. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσοι θα αποχωρούσαν ή όχι. Και το θέμα να ενισχυθεί το λειτουργικό σκέλος της όλα Επανειλημμένα το εξετάζουμε. Θα ήθελα να σας αναφέρω στην περίπτωση που γινόσαστε γενικό διευθυντή, ποια προθεσμία θα υπήρχε για μια τέτοια σε βάθο ε, μεταρρύθμιση και σε σχέση με τα εσωτερικά προβλήματα ε, και τις αντίπερα όχθη, ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστία. Εσεί μα δώσατε ω αναφορά ότι άλλοι διεθνείς οργανισμοί ότι έχουν χειρότερα ποσοστά ή αποτελέσματα από ότι η Όλαφ. Δεν μα παρηγορεί αυτό. Εσεί πώ θα αναλαμβάνατε ηγετικό ρόλο για να πάψει αυτό το πρόβλημα και για να είσαστε σημείο αναφορά όσον αφορά την εσωτερική πειθαρχία, διότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλη σημασία μέσο. Ευχαριστώ. Well, thank you guys. Ευχαριστώ. Μπορεί να γίνει η εξοικονόμηση πόρων στην όλαψη ό,τι αφορά το λειτουργικό της μέρος. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα ακριβής ε, για γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα με κατηγορήσουν ορισμένοι επικεφαλής ε, προϊστάμενοι τμήματων ότι προσπαθώ να πάρω τη δουλειά τους. Συγχωρήστε με λοιπόν αν δεν είμαι απόλυτα ακριβής. Υπάρχουν όμως ε, τομείς όπου μπορούν να γίνουν ε, οικονομίες και όπου θα πρέπει να μετατεθεί η προσοχή που, που στην εστιάζουμε. Πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένες συνέργειες στις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι υπεύθυνη για τα περιφερειακά ταμεία, τη γεωργία και τα τελωνία. Νομίζω ότι θα πρέπει να, αναδιοργανώσουμε διοργανώσουμε τον τομέα αυτό. Θα χρειαστούν 6 18 μήνες ε, στην Επιτροπή. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα σε ό,τι αφορά το θέμα της ηγεσία. Ε, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας θεωρώ ότι είχα αρκετά ηγετικό ρόλο στην Όλαβη για αρκετά χρόνια, όχι για μερικούς μήνες. Πιστεύω ότι το έκανα καλά, πιστεύω ότι συνέβαλα στο να ε, αντιμετωπίσουμε δύσκολους καιρούς. Και αυτό το βασίζω στην ανατροφοδότηση που έχω από όλες τις ομάδες και από όλες τις εθνικότητες μέσα στο γραφείο. Και πραγματικά με εξέπληξε το γεγονός ότι ε, επικροτήθηκαν τα, όσα είπα ακόμα και σε μια κηδεία, σε ένα επικίδιο. Είμαι πεπισμένος ότι θέτοντας το καλό παράδειγμα, επικοινωνώντας σωστά, έχοντας μια σωστή αντιμετώπιση όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες σχέσεις, θα καταφέρουμε να επιλύσουμε αυτά τα θέματα. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Θα έλεγα ότι οι προηγούμενοι δέκα μήνες ήταν αρκετά ήρεμοι. Συνάδελφος Ρενάουζερ. Ευχαριστώ Θέμα, για την πολιτική άσκηση επιρροής. Εσείς ο ίδιος μέσω των ε, εξουσιών θα εξαρτάστε από πολιτική απόφαση Βλέπετε άσκηση επιρροής πολιτικά ως πρόβλημα και κυρίως ε, θα με ενδιέφερε αν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί, αν πιστεύετε ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ήδη την άσκηση επιρροής την κρατούν σε ένα ελάχιστο ε, επίπεδο που θα ήταν αναγκαίο ή αν έχετε κάποιες ε, καινοτόμες προτάσεις πώς θα μπορούσε να μειωθεί η πολιτική επιρροή προς όφελος της διαφάνειας. Ευχαριστώ. Η απάντηση είναι διαφανειας απλή. Όχι. Όχι κύριε δεν βλέπω κανένα πρόβλημα με την άσκηση πολιτικά άσκηση επιρροής. Ποτέ δεν ασκήθηκε πολιτική επιρροή σε έρευνες. Τελείο. Τελείο και παύλα. Αυτή ήταν η απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Άιλετ για την ακρόαση αυτή και τον χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Allora, procediamo alla ultima audizione. Περνάμε στην τελευταία ακρόαση. κύριο Τζοβάνι Κέσλερ, επιτρέψτε μου να του δώσω το λόγο, υπενθυμίζοντας ότι έχει πέντε λεπτά καιρό για την παρουσίασή του. Παρακαλώ κύριε Κέσλερ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους σας. Θα ήθελα σύντομα να σας συστηθώ και να διατυπώσω ορισμένες σκέψεις σχετικά με την όλα. Είμαι εισαγγελέα και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου είχα την δυνατότητα και την ευκαιρία να εργαστώ σε διάφορους τομείς σε εντελώ διαφορετικό πλαίσιο και να αντιμετωπίσω μια σειρά από περιπτώσεις. Ως εισαγγελέα στην πόλη μου ήμουν επικεφαλής μιας έρευνας που ετέλειψε στην εξάρθρωση ενός δικτύου διαφθοράς όπου ενέχονται εργολήπτες και επιχειρηματίες και σε συνεργασία με τη γερμανική ε, και βρετανική αστυνομία καταφέραμε να αποκαλύψουμε εταιρείε offshore στα νησιά του Καναλιού και στο Λίχνεστάιν όπου διοχετεύονται τα παράνομα χρήματα από την αποτέλεσμα διαφθοράς. Ήταν λίγο δύσκολη η περίπτωση του Λίξτεστάιν. Σε κάθε περίπτωση στέφθηκε από επιτυχία η έρευνα αυτή. Πολλοί καταδικάστηκαν και πάρα πολλά χρήματα ανακτήθηκαν. Ως εισαγγελέας κατά τις μαφίες στην Σικηλία ήμουν ε, επικεφαλής μιας έρευνας για μια ε, οικογένεια της μαφίας. Συνεργάστηκα με μια ομάδα ερευνητών και καταφέραμε να καταδικαστούν πάνω από 100 άτομα μέλη της μαφίας. Περισσότερο από 100 μαφιόζοι άτομα που είχαν σχέση με διαφθορά, με εκβιασμούς, ακόμα και με δολοφονίες. Ως εισαγγελέα στο Μπολτζάνο, μια πόλη που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία και την Αυστρία, ήμουν επικεφαλής μιας έρευνας που αφορούσε μια πάτη κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με τις τελωνικές υπηρεσίες της Ιταλίας και της Γερμανίας καταφέραμε να αποκαλύψουμε μια Ιταλική εταιρεία και οι ιδιοκτήτες αυτής της εταιρείας καταδικάστηκαν. Η εταιρεία αυτή χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποστολή επισητιστική βοήθεια στην Αλβανία, δεν έφτασε βοήθεια και τα τρόφιμα κατέληγαν στην Ευρώπη. Στο τέλος καταφέραμε να καταδικαστούν τα άτομα αυτά και να ανακτήσουμε τα χρήματα. Τα χρήματα τα οποία είχαν παρανόμως. Κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής μου σε διεθνές επίπεδο ορίστηκα επικεφαλής της αποστολής σε παλήθευση στο πέδιο. Ήμουν επικεφαλής της, του αστυνομικού και δικαστικού τμήματος της αποστολής και συνεργάστηκα με πάνω από 300 άτομα. Οργάνωσα επίσης και διεύθυνα την πρώτη κοινή επιχείρηση στην Ιταλία κατά της παραχάραξης, της παραποίησης και εστίασα την προσοχή μου στην Φλωρεντία για πρώτη φορά όλη η Ιταλική αστυνομία, τα τελωνία, ακόμα και η δημοτική αστυνομία και μέχρι τον ε, ε, τους αστυνομικούς της πόλης πήραν μέρος στην επιχείρηση αυτή η οποία οδήγησε στην κατάσχεση μιας σειράς παραποιημένων αγαθών που κατασκευάζονται σε παράνομα εργαστήρια και βεβαίως συνελήφθησαν και πάρα πολλά άτομα. Και αυτό βεβαίω, σε αυτό δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη έκταση στον τύπο και επενέργησε και αποτρεπτικά σε ό,τι αφορά τον τομέα της παραποίηση που πλήττει όχι μόνο την Ιταλία αλλά και όλη την Ευρώπη. Δύο λόγια για την Όλαφ. Θα αφιερώσω όλες μου τις ενέργειες στον τομέα της ανεξαρτησίας, της ενότητας και της αποτελεσματικότητας. Η Όλαφα χωρίς ανεξαρτησία δεν μπορεί να κάνει έρευνες, δεν έχει νόημα, δεν έχει χρησιμότητα. Είναι εύκολο να προσανατολίσω όλες μου τις δράσεις και τις δράσεις της Όλαφα προς την ανεξαρτησία γιατί αποτελεί μέρος της κουλτούρας μου, είμαι εισαγγελέα. Ενότητα μετά από τόσες εντάσεις και τόσες διαφορές η Όλαφ χρειάζεται ενότητα. Μπορώ να εξασφαλίσω την ενότητα, είμαι εκτός της Όλαφ και δεν έχω κάποια εσωτερική δέσμευση, δεν ανήκω σε κάποια ομάδα, δεν χρειάζεται να προασπίσω οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στο παρελθόν. Αποτελεσματικότητα. Θα μιλήσω για την αποτελεσματικότητα μετά από τις ερωτήσεις που θα θέσατε. Ευχαριστώ κύριε Γκρέσον. Κυρία Γκρέσλε πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κέσλερ, είχα μεγάλη, ας το πω προσπάθεια που κατέβαλα μαζί σας, περισσότερο από κάθε άλλον υποψήφιο. Έχω την εντύπωση ότι είσαστε γενικόλογος περισσότερο από τους άλλους. Θα ήθελα πιο χειροπιαστά, πιο εξειδικευμένα να αναφέρω. Βρίσκεται πέρα από δέκα χρόνια η δικαστική σας πείρα, η εμπειρία μετά γίνατε πολιτικός. Θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζουμε ποια είναι η πείρα σας από τον πολιτικό τομέα, τι θα συνεισφέρετε στην Όλαφ σχετικά και θα πρέπει να μας πείτε χειροπιαστά ποιες δραστηριότητες θέλετε να μειώσετε όταν περισσότεροι θα αφιερωθούν ως στελέχη στις ερευνητικές δραστηριότητες. Από πού θα αντλήσετε αυτά τα στελέχη, αυτό το προσωπικό. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει εν τω μεταξύ είπατε non-essential υπηρεσίες υπάρχουν, μη ουσιώδεις υπηρεσίες στην Όλαφ. Ποιε είναι αυτές οι μη ουσιώδεις υπηρεσίες. Ε, ε, Έχω πολιτική εμπειρία, αλλά είμαι πάντοτε εισαγγελέα. Και όσον αφορά την πολιτική, θέλω να πω ότι και τις γνώσεις μου ως εισαγγελέο ε, τις προσέφερα στην πολιτική. Δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου και θεωρούμε ως ένας εισαγγελέα που έχει γνώση της πολιτικής και στην πολιτική μου δέσμευση προσέφερα την κουλτούρα mm. του κανόνα δικαίου στο κοινοβούλια και έχω αφοσιωθεί για τις επιτροπές ε, έρευνας, ε, εξεταστικές επιτροπές ε, στον τομέα, το, στην Επιτροπή Δικαιοσύνης και Νομικών Υποθέσεων. Τώρα, για το δεύτερο σκέλος της ερώτησή σας, θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία στις έρευνες για, και να δώσουμε περισσότερους ανθρώπινους και πόρους σε αυτές τις έρευνες τι μπορεί κανείς να μειώσει για να αυξήσει αυτό το τομέα. Μίλησα για την αρχή της επικουρικότητας, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται και στις δραστηριότητες της Όλαφ. Το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούν να βελτιωθούν πιο αποτελεσματικά από τα θεσμικά μας όργανα θα πρέπει να περιοριστούν από την Όλαφ. Για παράδειγμα, η οικονομική παρακολούθηση, η χρηματοοικονομική παρακολούθηση. Πιστεύω εγώ προσωπικά ότι στην Όλαφ υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, περισσότερα από 100, που ασχολούνται με την χρηματοοικονομική παρακολούθηση της έρευνας. Ενώ αυτό το σκέλος μπορεί να καλυφθεί με την ίδια αποτελεσματικότητα από γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής, για παράδειγμα. Επίσης, η συλλογή στρατηγικών πληροφοριών, που είναι κάτι το σημαντικό βέβαια, αλλά πιστεύω πάλι ότι πολλοί πόροι προσανατολίζονται, ανθρώπινοι πόροι, προσανατολίζονται προς αυτήν την κατεύθυνση και θα μπορούσαν καλύτερα να χρησιμοποιηθούν ή μέρος αυτών τουλάχιστον για τις έρευνες που εξάγονται. Ευχαριστώ. Γκάιε, παρακαλώ. Κύριε Κέσλερ, καλώς ήρθατε θερμά στην Επιτροπή μας. Εντυπωσιάστηκα από αυτά που διάβασα για σας και αποκόμισα την εντύπωση, πιστεύω, ότι κανείς σε σχέση με σας δεν έχει, πώς να το πω, δεν ταιριάζει η περιγραφή σε αυτόν όπως ε, η προκήρυξη για τον υποψήφιο Γενικό Διευθυντή που ταιριάζει τόσο σε εσά. Η Όλαφ είναι μια ειδική υπηρεσία. Εργάζεται όχι μόνο σε ένα διεθνέ παγκόσμιο περιβάλλον, αλλά έχει και ένα ειδικό, ιδιαίτερο ρόλο όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μεταξύ των θεσμικών οργάνων και αναμεταξύ της. Είναι σαφές ότι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εργαστήκατε και, έχετε, ε, και υπάρχουν κάποια προτερήματα στις πληροφορίες σχετικά. Θα με ενδιαφέρει να ξέρουμε ποια πείρα έχετε από τη διεθνή σας εμπειρία που θα σας συνεισέφερε να είσαστε καλό γενικός διευθυντής της Όλαφ. Yeah, uh, I think they... Νομίζω ότι ο διευθυντής τη Όλαφ φυσικά θα πρέπει να έχει πείρα όσον αφορά τις έρευνες και τις ανακρίσεις που γίνονται, εφόσον είμαστε ένας οργανισμός ερευνών, θα πρέπει να έχει ε, διοικητικές ικανότητες και εμπειρία, εφόσον θα διοικεί πάνω από 500 άτομα και επίσης θα πρέπει να ελέγχει τον ετήσιο προπολογισμό, αλλά όπως είπατε ο Διευθυντής τη Όλαφ θα πρέπει επίσης να έχει και πολιτική εμπειρία, επειδή η Όλαφ είναι ένας οργανισμό που διαμορφώνει και πολιτική, μαζί με του, τους άλλους ενδιαφερόμενους. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εν ώψη της μεταρρύθμισης της Όλαφ, την οποία ε, συζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο και με την προοπτική ε, της βελτίωσης του ρόλου, της αναβάθμισης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Συνηγόρου, νομίζω ότι ο ρόλος ε, του Διευθυντή της Όλαφ είναι πολύ σημαντικός επειδή μπορεί να συμβάλλει, να δίνει τις συμβουλές του και η εμπειρία που έχω και στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών και συνελεύσεων και στον πολιτικό κόσμο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα με βοηθήσουν να είμαι όχι μόνο ένα άτομο το οποίο θα διεξάγει τις έρευνες, ένα στοιχείο της όλα αλλά θα μπορώ να συνεργάζομαι στενά με το Κοινοβούλιο, με την Επιτροπή, σε αυτή τη διαδικασία για την ε, διαμόρφωση της μεταρρύθμισης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Γκρέσλε, ακριβώς. Αυτά σε σχέση με την Ιταλία. Επανέρχομαι. Στην παρουσίασή σας, στα γραπτά σας έγγραφα που έχουμε, κάνετε λόγο για irrelevant cases, άσχετες περιπτώσεις. Irrelevant cases, δηλαδή άσχετες ε, περιπτώσεις στις οποίες ε, κάνει έρευνες η Όλαφ. Παλαιό πρόβλημα αυτό και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο ειλικρινείς αναμεταξύ μας από ό,τι μέχρι τώρα στο ερώτημα πότε βλέπουμε ότι κάτι είναι άσχετη περίπτωση πότε δια... μπορεί να υπάρξει διάγνωση ότι αξίζει να γίνει έρευνα ή όχι το ερώτημα είναι όταν υπάρχει επαρκής υποψία πώς πρέπει να αντιμετωπίζει τέτοιες περιπτώσεις ε, η Όλαφ ήταν πάντα πολιτική του σώματος τέτοιου είδους περιπτώσεις ε, να αντιμετωπίζονται και να αποφεύγονται. Πώς ξέρουμε όμως ε, ότι μια τέτοια περίπτωση είναι άσχετη. Ποιες αλλαγές μέσα στην όλα θεωρείτε ότι είναι αναγκαίες ώστε να μπορέσουν πιο γοργά να διαπιστώνονται τέτοιου είδους άσχετες περιπτώσεις. Όπως είπατε, είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα γιατί αφορά την αποτελεσματικότητα την, ε, και ε, την διαφάνεια. Υπάρχει κάτι που αρχικά φαίνεται να είναι άσχετο, ενώ αποδεικνύεται ότι δεν είναι καθόλου άσχετο. Πώς μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι όμως Διαφορετικά η Όλαφ θα επικεντρώνεται μόνο σε περιπτώσεις ελάσσονος σημασίας. Καταρχάς χρειάζεται ένας κανονισμός. Δεν μπορεί αυτό να αφαιθεί στη διακριτική ευχέρεια της, ε, του διευθυντή της Όλαφ ή στη διακριτική ευχέρεια οποιοδήποτε καταρχάς. Πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η de πολιτική η οποία εφαρμόστηκε τουλάχιστον σε μια αρχική φάση η οποία εστιάζεται πρωτίστως σε ένα προσωπικό, ε, ποσοτικό με κατόφλι. Αυτός είναι ένας στόχος που θα μπορούσε να βοηθήσει. Κατά την άποψή μου όμως δεν είναι το μοναδικό σημείο αναφοράς για να αναγνωρίσει κανείς ε, τη σχετικότητα μιας περίπτωσης το δεύτερο σημαντικό στοιχείο για να καθορίσει κανείς αν κάτι είναι σχετικό ή άσχετο για την Όλαφ, για την Όλαφ, τον υπογραμμίζω, όχι αντικειμενική σχετικότητα, είναι η χρήση της αρχής της επικουρικότητας, που σημαίνει ότι αν υπάρχει κάποια, κάποιος άλλος φορέας, όπως είναι για παράδειγμα, που μπορεί να κάνει τη δουλειά, τότε είναι άσχετη θα το λέγαμε περίπτωση για την Όλαφ και η Όλαφ μπορεί να το ε, προωθήσει στην ΆΙΤΟ και να παρακολουθεί. Αλλά μία μικρή περίπτωση όπου η ΙΔΟΚ η δεν έχει αρμοδιότητες, τότε αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει να για αυτές τις περιπτώσεις ε, θα πρέπει να επιλαμβάνεται η Όλαφ μόνο ότι το ποσοτικό κατόφλι είναι αρκετά χαμηλό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υποψήφιε, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υποψήφι, Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής σας ενημερωθήκαμε για την πείρα που έχετε στον ε, τομέα της εισαγγελίας αλλά και για άλλους ε, τομείς. Δεν μιλήσατε όμως για το όραμά σας. Πώς τη βλέπετε την Όλαβα. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα αυτές τις μέρες. Εγώ είμαι καινούριο μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω, ξέρω όμως ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός στο προσωπικό της Όλαφα. Εσείς θα ηγηθείτε αυτού του φορέα και θα κληθείτε να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα. όταν βρεθείτε αντιμέτωποι με την δυσαρέσκεια του προσωπικού. Από την άλλη πλευρά, ενδεχομένω υπάρχουν προβλήματα που αφορούν την επικοινωνία, τις σχέσεις με τις χώρες μέλη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο σύστημα έτσι ώστε οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μελών και της Όλαφ να είναι καλές. Η Όλαφ όσο δομή δεν ξέρει πώς θα πρέπει να δράσουν οι χώρες μέλη. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των χωρών μελών, τι θα πρέπει να κάνουν στο δικό τους επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση των συγκρούσεων στο εσωτερικό της Όλαφ. Το δεύτερο ερώτημα να μου πείτε τι θα πρέπει να αλλάξει στις σχέσεις μεταξύ της Όλαφ και των χωρών μελών έτσι ώστε η διαδικασία έτσι ώστε η διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ. As αφορά την εσωτερική κατάσταση, ναι. Άλλωστε, στο εξωτερικό φαινόταν ότι υπάρχει κάποια διχασμός, ορισμένες ομάδες συγκρουόμενες ε, στην Όλαφ. Αλλά βρίσκομαι σε καλή θέση, επειδή εγώ δεν ανήκω σε κανένα μια από αυτές τις ομάδες. Η πολιτική μου λοιπόν θα ήταν εξή. Συμμετοχή όλων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα όλα τα ανώτερα στελέχη, όλο το προσωπικό να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, δηλαδή να μπορούν όλοι να διατυπώνουν τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και να έχουν το δικαίωμα να συζητούνται όλα αυτά με διαφάνεια. Συνεπώς, δύο λέξει: Συμμετοχή και διαφάνεια των αποφάσεων για να εξασφαλιστεί η σωστή βάση για να λαμβάνονται αποφάσεις με γνώμονα τα συμφέροντα και τις προτάσεις των υπαλλήλων. Αυτή τη στιγμή αποφασιστεί ένα θέμα με συμμετοχικό και διαφανή τρόπο, θα πρέπει όλοι να σεβαστούν τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και να μην υπάρχουν κρυφές ατζέντε, να μην υπάρχει προσφυγή προς τα έξω. Αυτό δεν θα γίνει δεκτό. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Αναζητείτε βοήθεια ή αναζητούνται συμμαχίες απ' έξω. Αυτή τη στιγμή έχει ληφθεί μία απόφαση με τρόπο συμμετοχικό και διαφανή. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα στροφής προς τα έξω. Δεν θα επιτραπεί αυτό. Ως προς τις σχέσεις με τα κράτη-μέλη, είναι διαφορετικές οι σχέσεις ανάλογα με τα κράτη-μέλη και υπάρχουν πραγματικά μερικές φορές προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με δύο τρόπους. Από την πλευρά της Όλαφ, και νομίζω ότι ο νέος μας κανονισμός, χρειάζεται ένας νέος κανονισμός νομίζω, και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μεταρρύθμιση του κανονισμού της Όλαφ. Στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου του 2008 δεν έχει ληφθεί υπόψη, ναι, αλλά δεν έχει ληφθεί παρκώς υπόψη στην πρόταση της Επιτροπής. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα σημείο αναφορά από το κάθε κράτο μέλο όσον αφορά τι σχέσει με την Όλαφ. Υπάρχουν περιοδικέ αναφορέ των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη σχετικά με τι έρευνε τη Όλαφ. Αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Και τρίτον, ένα νέο κανονισμό για την αποτελεσματικότητα των τεκμηρίων που έχει βρει η έρευνα της Όλαφ. Ο κ. Χατζημαρκάκης. κύριε Κέσλερ, η παρουσίασή σας μου άρεσε ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα η όρη ανεξαρτησία, ενότητα, αποτελεσματικότητα. Ξεκινώ με την αποτελεσματικότητα και προσθέτω τη φωνή μου στην ερώτηση του συναδέλφου Μπάτσιτης στο θέμα των σχέσεων με τα κράτη-μέλη, με κράτη-μέλη, σε σχέση με αυτά δηλαδή. Πολλές από τις περιπτώσεις συναποτελούνται από τρία, τέσσερα, και πάνω από πέντε χρόνια στην Όλαφ. Ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Δυστυχώς οι σχέσεις με τα κράτη-μέλη είναι ιδιαίτερα αποφασιστικές. Διότι πολύ συχνά η παρακολούθηση ερευνητικά γίνεται από τα κράτη-μέλη μετά από εσά. Πώς θέλετε σε αυτό το σημείο τη σύνμηση των ε, διοριών και των προθεσμιών. Τι θα κάνετε προσωπικά γι' αυτό. Ε, Υπάρχουν δύο λόγοι που με κάνουν να ανησυχώ για την παρούσα κατάσταση της όλα και αυτό ε, σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα και την έλλειψη αποτελεσμάτων, αποτελεσμάτων ε, δικαστικών στις χώρες μέλη. Σε ένα μισή λεπτό θα πρέπει να σας τα πω όλα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κινηθούμε με δύο τρόπους μέσα στην Όλαβα. Πέρα από το θέμα της μεταρρύθμισης του κανονισμού, ένα θέμα που ήδη έθιξα, θα πρέπει να ζητήσουμε την συνδρομή του δικαστικού προσωπικού της Όλαφ στις έρευνες αυτές σε μία πρώιμη φάση, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα. Ε, μπλέκονται μόνο στο τέλος των ε, ερευνών ή στη συνέχεια. Η πρώιμη συμμετοχή τους, η έγκαιρη συμμετοχή τους θα και δύο αποτελέσματα. Καταρχάς θα μπορέσουν να επηρεάσουν περισσότερο τα πράγματα ή να επηρεάσουν τις εθνικές δικαστικές αρχές ε, γιατί θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι έρευνε τη Όλαφ στρέφονται και προ τι εθνικέ δικαστικέ αρχέ. Αν προέρχονται από έναν συνάδελφο, από έναν εισαγγελέα, ο εισαγγελέα ξέρει πώς οι συναδελφοί του σε μια χώρα μέλο λειτουργούν και μπορεί να επηρεάσει περισσότερο τα πράγματα έχοντα κατά νου την επίτευξη ενό συγκεκριμένου αποτελέσματο. Δεύτερον, τα συμβάλλουμε στο να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των ατόμων που μπλέκονται στις έρευνες και αυτό χρησιμοποιώντας και δικαστικό προσωπικό και ζητώντας τους να πάρουν μέρος στις έρευνες. Η κουλτούρα που έχουν είναι διαφορετική από αυτή της αστυνομίας. Αυτός είναι ένας τρόπος. Το δεύτερο που θα ήθελα να αναφέρω είναι εκεί που είναι δυνατόν αλλά θα έλεγα σε όλες τις περιπτώσεις να ζητήσουμε τη συνδρομή της εθνικής αστυνομίας και των δικαστικών αρχών στις έρευνες της Όλαφα. Όχι μόνο να τους δίνουμε τα αποτελέσματα των ερευνών, μια έρευνα για την οποία δεν γνωρίζουν τίποτα. Εάν έχουν μία έγκαιρη εμπλοκή στι ε, έρευνες, ακόμα και τα στατιστικά δεδομένα μας λένε ότι οι επιτυχίε είναι πολύ περισσότερες στι χώρες μέλη από ότι όταν οι δικαστικές, οι αστυνομικές αρχές καλούνται να πάρουν μέρος σε μία μετέπειτα φάση. Συναδέλφο Καλώς ήρθατε. Πρώτα απ' όλα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ ανταπαντά ο υποψήφιος. Καλώς ήρθατε λοιπόν, κύριε Κέσλε. Μάλιστα. Θα ήθελα να δώσω συνέχεια σε αυτό το σημείο για τη συνεργασία με άλλους Κάνατε λόγο για συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Όμω, κάποιοι υποψήφοι πριν από εσά μίλησαν και για πιθανή συνεργασία με άλλου οργανισμού όπω τη Europol, τη Eurojust κτλ. Ερώτημα προ εμά. Νομίζετε ότι υπάρχει κάποιο δυναμικό για τέτοια συνεργασία. Σε ποιο βαθμό η Όλαφ θα μπορούσε να συνεργαστεί με οργανώσει όπω τη Eurojust, η Europol, συμπληρώνεται και με την δική σα πείρα. Θα ήταν καλή ιδέα αυτή. Ε, of course, ε, Βεβαίως, η Όλαφ πρέπει να συνεργάζεται με τους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την αντιμετώπιση των ίδιων θεμάτων, δηλαδή με τη Europol και τη Eurojust. Αλλά είναι διαφορετικό από το να συνεργάζεσαι με τις εθνικές αστυνομικές αρχές ή τις δικαστικές αρχές. Ήδη υπάρχει μια τεχνική πρακτική συμφωνία μεταξύ Eurojust και Olaf και θεωρώ σημαντικό όχι απλά να συνεργάζεται κανείς ε, πάνω στο ίδιο θέμα, στην ίδια έρευνα, αλλά και σε αυτά τα οποία ανέφερα προηγουμένως που συνοψίζονται στη λέξη επικουρικότητα. Δηλαδή, να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Μπορούμε να δίνουμε πληροφορίες στην Eurojust και η Eurojust το ίδιο με εμά, συνεπώς χρειάζεται συνεργασία μεταξύ μας. αλλά όχι απαραίτητα επιχειρησιακή συνεργασία πάνω στο ίδιο θέμα, διότι τελικά θα υπάρξουν επικαλύψεις ε, και χάσιμο πόρων. Αυτό το οποίο μας χρειάζεται αντιθέτω είναι συνεργασία στις ίδιες υποθέσεις μεταξύ των ερευνητών της Όλαφ και των εθνικών ερευνητών. Ευχαριστώ. Κύριε Ανδρέασεν. Κύριε Κέσλερ, όταν μας παρουσιάσατε την υποψηφιότητά σας, υπογραμμίσατε τις πολιτικές σας ικανότητες. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κατά πόσον πιστεύετε ότι αυτές οι πολιτικές σας ε, ικανότητες και η πείρα είναι σημαντικές για το ρόλο του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ. Δεύτερον, ε, μου φάνηκε ότι δεν δώσατε τόσο πολύ μεγάλη σημασία στη στρατηγική πληροφόρηση. Μπορείτε να μου πείτε ποια μέτρα προτείνετε ω γενικό Διευθυντής τη Όλαφ για να βελτιώσετε την, απο, ε, την αποτελεσματικότητα στην διαπίστωση, την ανείχνευση της απάτης. Θα αρχίσω με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Σύμφωνα με τις στατιστικές, πάρα πάρα πολύ λίγες υποθέσεις τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν από την στρατηγική πληροφόρηση. Όταν λέω πολύ πολύ λίγες, ίσως όχι περισσότερες από 4 ή 5 ετησίως, ε, πάνω σε 3-4 χιλιάδες ετησίως. Λοιπόν, η στρατηγική τεσσερις χιλιαδες ετησιως λοιπον είναι μεν σημαντική, αλλά όχι ως χρήσιμη πηγή πληροφοριών για να ξεκινήσει κανείς μια έρευνα. Είναι χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες για την διαμόρφωση της πολιτικής στην Όλαφ, ώστε να προσανατολίζεται όχι τόσο η Όλαφ οι έρευνές της, αλλά η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών οργάνων και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποτρέπεται η απάτη. Αλλά δεν χρησιμεύει ε, στην καθαυτό έρευνα. Δεν θέλω να μειώσω τη σημασία των στρατηγικών πληροφοριών, αλλά αν θέλω να βελτιωθεί το επιχειρησιακό σκέλος της Όλαφ, που είναι η δουλειά μας, η βασική δουλειά των ερευνών, της ανάκρισης. Και αν γνωρίζω ότι το σύνολο των ανθρωπίνων και υλικών πόρων είναι δεδομένο, τότε θα πρέπει να μεταθέσω πόρους από τον ένα κλάδο στον άλλον. Και ένας κλάδος, ένας τομέας, όπου βαθμιαία θα αφαιρούσα πόρους, είναι η στρατηγική πληροφόρηση. Δεν θα το διέλει αυτό το τομέα, αλλά θα τον μείωνα. Διότι θέλω να εστιάσω περισσότερο στην γενική πληροφόρηση. Τώρα, σχετικά με την πολιτική πλευρά τι εμπειρίας μου, την πολιτική μου διάσταση αν θέλετε, ήμουν, υπήρξα και είμαι ε, εισαγγελέα, υπήρξα και εισαγγελέα ε, στο Κοινοβούλιο και το έργο το οποίο επετέλεσα στο Κοινοβούλιο είχε ως βάση το εισαγγελικό μου καθήκον και το ίδιο θα πράξω στην Όλαφ γνωρίζοντας ότι αν είμαι διευθυντής της Όλαφ, το να είμαι μόνον ερευνητή ή εισαγγελέας, αυτό δεν αρκεί. Θα γνωρίζω το έργο αυτών των δύο αξιωμάτων, αλλά ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ θα πρέπει να γνωρίζει πώς θα αντιμετωπίζει θέματα που έχουν σχέση με τους βουλευτές, ευρωβουλευτές και τα πολιτικά θεσμικά όργανα. Συνάδελφος Πατρίση. Η Όλαφ είναι μια ε, ε, ερευνητική υπηρεσία, τη οποία ο Γενικό Διευθυντή θα πρέπει να είναι και να φαίνεται ε, ανεξάρτητος, χωρίς να υπόκειται σε επηρεασμούς πολιτικούς. Τρεις ερωτήσεις. Δεν πιστεύετε ότι το να είναι κανείς πολιτικός θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε εσά και στην Όλαφα όταν οριστείτε γενικός διευθυντής. Δεύτερον, πώς θα μπορέσετε να προσπίσετε το γραφείο και τις έρευνες από τις ε, κατηγορίες ότι σας υποκινούν πολιτικά αίτια. Τρίτον, τι σχέση θα έχετε ως πολιτικός με τους επιτρόπους της Επιτροπής και με το Κοινοβούλιο ως ανώτατος αξιωματούχος. Well, yeah, it is true, as ναι. Αληθεύει όπως λέτε ότι η ανεξαρτησία έχει τεράστια σημασία όπως είπατε. Και δεν αρκεί να είναι κανείς ανεξάρτητος για ένα θεσμικό όργανο. Πρέπει και να φαίνεται και να δείχνει ανεξάρτητος, σίγουρα. Εγώ είμαι πολιτικός άνδρας, ναι. Είμαι ένας δημόσιος κατηγόρος εισαγγελέας που ασχολείται με την πολιτική εδώ και κάποιο διάστημα. Δεν είμαι όμως σταδιοδρομίας πολιτικός, επαγγελματίας πολιτικός. Όταν ήμουνα στην Βουλή δεν ήμουνα μέλος κανενός κόμματος. Ήμουνα ένας εισαγγελέα που ασχολήθηκε με τα πολιτικά. Ήμουνα το μόνο μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας στο κοινοβούλιο μας χωρίς να ανήκω σε κάποιο κόμμα. Και γνωρίζετε τι σημαίνει να είναι κανείς ανεξάρτητος όσον αφορά ένα κόμμα. Και πάντα έτσι με έβλεπαν και πάντα ήμουν αμερόληπτος στην πολιτική μου δράση, ακόμα και τώρα. ήμουν πιο ε, δημοφιλής και με τις περισσότερες ψήφους στον, ε, στην λίστα μου και σε σχέση και με την ε, κυβέρνηση, την περιφερειακή κυβέρνηση, ήμουν όμως μέλος της, νομοθετικ... του νομοθετικού, της νομοθετικής βουλής. Ήμουν αμερόληπτος και είχα ψήφους που με υποστήριξαν και από την αντιπολίτευση δεν ήμουν και ποτέ δεν θεωρήθηκα ένας μεροληπτικός κομματικός πολιτικός ή ένας τυπικός κομματικός πολιτικός άνδρας, διότι δεν ήμουν τέτοιος. Δεύτερον, πώς θα μπορούσα να υπερασπιστώ την Όλαφ από τέτοιου είδους κατηγορίες πολιτικής μεροληψίας. Είμαι συνηθισμένος σε αυτά τα θέματα. Όταν ήμουν εισαγγελέα, καθόλου δεν είχα αναμειχθεί σε πολιτικά θέματα. Δεν είχα ούτε και πολιτική πείρα η προηγούμενη σταδιοδρομία. Πολλές φορές με κατηγόρησαν ότι είχα πολιτικές μεροληψίες ή πολιτικές κατευθύνσεις ε, σε σχέση με κάποιες επαφές. Ε, κάποιοι με κατηγορούσαν ότι ήμουν αριστερός ε, όσον αφορά τους δεξιούς. Αργότερα λόγω κάποιων επαφών με άλλους κατηγορήθηκα ότι ήμουνα δεξιόστροφος, δεξιός πολιτικός. Είμαι συνηθισμένος να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου πρέπει να πω ή το θεσμικό όργανο που εκπροσωπώ σε σχέση με τέτοιες κατηγορίες λόγω της συμπεριφοράς μου της ίδιας και για τα, από τα αποτελέσματα που επινηχάνω. Ως επικεφαλής της Όλαφ πρέπει να μπορεί να συνεργάζεται κανείς πολύ στενά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Όλαφ είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όταν έχει η ώρα της πολιτικής, ε, του πολιτικού σχεδιασμού πρέπει να συνεργάζεται κανείς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή ιδιαίτερα που θεωρώ ότι είναι υπαριθμόν ένα ε, υπέρμαχος ε, των αρμοδιοτήτων και της ανεξαρτησίας από πλευρά των συμφερόντων των πολιτών της Ευρώπης που εκπροσωπείται. Ο, ο Κύριε Χέιζελ, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε δύο σημεία που αναφέρατε με θαυμάσιο τρόπο στην αρχή. Το θέμα της ανεξαρτησίας πρωτίστως. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και μία άλλη έννοια την ανεξαρτησία όχι μόνο από την πολιτική αλλά από ισχυρές δυνάμεις που επηρεάζουν τα πράγματα πολύ περισσότερο. Επηρεάζουν τη δυνατότητα ελέγχου που έχετε και πολέμηση της απάτης στην Ευρώπη. Μιλάμε για λόμπι και μερικές φορές για λόμπι αρκετά σκοτεινά, αδιαφανή. Εμένα με ενδιαφέρει ένα διευθυντή τη Όλα που είναι αναπόλυτα ανεξάρτητο από αυτή την άποψη. Επειδή γνωρίζω τη δράση σα στην Ιταλία Πραγματικά αναρωτιέμαι πώ θα μπορούσατε αυτή την πείρα σα να τη θέσετε στην υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Δεύτερο θέμα, το θέμα τη αποτελεσματικότητα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα και αυτό με τη σειρά του που αφορά την υπάρχουσα δομή τη Όλαφ και του τρόπου με τον οποίο σκέφτεστε με βάση τι εμπειρίε που αποκτήσατε σε διεθνέ πλαίσιο να την αναδιαρθρώσετε σε μια σχέση συνεργασία με το Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Ευχαριστώ. Το πρώτο μέρος της ερώτησής σας. Συμφωνώ μαζί σας. Με απασχολεί περισσότερο, με βάση τα όσα έχω βιώσει μέχρι τώρα, ο τομέας που αφορά τα διαφανή, τα συγκαλυμμένα συμφέροντα. Η πολιτική είναι αρκετά διαφανή τις περισσότερες φορές αλλά είναι δύσκολο να δει κανεί τις επιρροές που προέρχονται από σκοτεινά συμφέροντα. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει πολιτική πείρα για να φεθεί, να επηρεαστεί από ε, συγκαλυμμένα οικονομικά συμφέροντα. Γι' αυτό το λόγο είπα ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στην όλα έτσι ώστε να δίνει κανείς και την εντύπωση ανεξάρτητου. Χρειάζεται βεβαίως και ε, ένας σαφής κανονισμός ε, να μην αφήνεται μεγάλη διακριτική ευχέρεια στην Όλαφ και στο Διευθυντή. ω διευθυντή τη Όλαφ θα ζητήσω να έχω έναν καλύτερο, ένα σαφέστερο κανονισμό που θα συνταχθεί από το Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή Ο κύριος Σρέσλε αναφέρθηκε προηγουμένως στο θέμα της πολιτικής de ε, για να ξέρουμε πότε και πώς ενημερώνουμε άτομα και φορείς σχετικά με τις διεξαγόμενες έρευνες. Κάτι που θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση της διαφάνειας και σε τελευταία ανάλυση και της εικόνας ε, ε, ανεξαρτησίας που προβάλλει. Σόντεργκερ. Κύριε Κέσλερ, νομίζω ότι... Θα μιλήσω αγγλικά. Προσέξτε. Την τελευταία φορά όταν συνεργαστήκαμε, είσαστε προεδρεύων επικεφαλής της ε, αποστολής παρατηρητών στα Ηνωμένα, ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου και μπορώ να πω ότι μπορείτε, μπορεί να αναλαμβάνετε πρωτοβουλία και σε μια πολυπολιτική αντιπροσωπεία. Μια ερώτηση θα ήθελα να διατυπώσω στις σχέσεις με τα κράτη-μέλη αλλά ήδη υπήρξε τοποθέτηση σχετικά και θα ήθελα να εμβαθύνετε σε κάτι το οποίο μόλις προαναφέρατε, τις σχέσεις με το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν είχατε την δυνατότητα να εκφράσετε κάποιες σκέψεις, αν κάποιες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν ή όχι, όσον αφορά το έργο της Όλαφ και σε επαφή με το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό θα ήθελα να μας πείτε περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στην κοινή μας εμπειρία στις Ηνωμένε Πολιτείε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών γιατί μου τέθηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική μου θέση. Είναι πολιτική, δεν είναι κομματική ε, θέση. Η αποστολή στις Ηνωμένε Πολιτείες κατά τη διάρκεια των πολιτικών εκλογών, των εκλογών στέθηκε από επιτυχία. Ε, στην αρχή υπήρχε μεγάλο σκεπτικισμό από πλευρά των Αμερικανικών αρχών και των ΜΜΕ, αλλά πραγματικά τα καταφέραμε όχι μόνο να κάνουμε μια αναφορά, μια έκθεση για τις ε, εκλογές, αλλά να αξιολογήσουμε την υπάρχουσα εκλογική νομοθεσία και να διατυπώσουμε προτάσεις μεταρρυθμιστικές τις οποίες προωθήσαμε και συζητήσαμε στο Αμερικανικό κάνει ε, Κογκρέσιο και το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτές είναι διεθνείς εμπειρίες που είναι και πολιτικές εμπειρίες που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αυτό ήταν ε, μόνο ένα παράδειγμα. Υπήρξαν και άλλες παρεμφερείς αποστολές σε άλλες χώρες και ασχολήθηκαν όχι μόνο στο κράτος δικαίου και στην εκλογική διαδικασία που ήταν σημαντική, αλλά εστιάστηκαν και στη διαδικασία μεταρρύθμισης ε, των εκλογών. Το ίδιο, ο ε, την ίδια συνεργασία θα επιθυμούσα να έχω και εδώ ως διευθυντής της Όλαβ και πιστεύω ότι αυτή μου η εμπειρία θα με βοηθήσει ιδιαίτερα στο να συμβάλλω όχι μόνο σαν ομομαθής ως δικηγόρος αλλά και ως πολιτικό όν, Να συμβάλλω δηλαδή στη μεταρρύθμιση της ε, Όλαφ σε επίπεδο κανονισμού. Κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και άλλα και αλλαγή των σχέσεων μεταξύ της Όλαφ και των χωρών μελών σε επίπεδο δικαστικών και αστυνομικών αρχών. Γιατί αυτό θα με βοηθήσει το να συμβάλλω στις προσπάθειες που καταβάλλονται και που αφορούν το Γενικό Εισαγγελέα. Ευχαριστώ. Τελείωσε η τελευταία ακρόαση. Ευχαριστούμε τον κύριο Κέσλερ. Ε, Ωραία. Θα συναντηθούμε στις 9 Νοεμβρίου και θα αποφασίσουμε για το διευθυντή της Όλβες 12 θα φύγει ένα λεωφορείο για το αεροδρόμιο. Στι 12, εκεί που είναι η σοφέρ. Σπινέλη Μπίλτη. Κύριο Σπινέλη. Τι να το πω, yes.